την περιοχή πέρα από τα Καρπάδια όπου καταστράφηκαν ε, μοναστήρια και για τις εκλογές ε, θα έπρεπε να διευκρινίσει τη θέση της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε ο συνάδελφος Σαλεύσκη τώρα. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική εβδομάδα για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας ήταν μια πάρα πολύ επικοδομητική εβδομάδα από αυτή την